Έχουμε μια ερώτηση που το Γιατί για αυτές τις επιχειρήσεις, αυτά που έγιναν στην Ουγγαρία. Και ιδίω η καταπλήρωση της πειρατείας. Εδώ και κάποιους μήνες κάναμε μια περιοδία στην περιοχή, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία κάποιων χωρών και της Κένια και των Σεϊχελών και άλλων ε, όσον αφορά την δικαστική συνεργασία για την αντιμετώπιση της ε, πειρατείας. Πρώτα για κάποιες προσπάθειες, ε, οι οποίες ακόμη δεν έχουν δώσει αποτελέσματα, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Αυτό αναφέρθηκε. Πώς έχουν τα πράγματα. Έχουμε τον κύριο Λάγκ, του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, τα αναφερόμενα για το ότι θα πρέπει να, να υπάρξει συνεργασία στην Άουσα, αλλά και στην ε, Βουδαπέστη. Επίσης ε, υπήρξε συζήτηση και για πετε μας πώς προχωρήσαμε όσον αφορά τη σχέση με τις χώρες αυτές. Και αυτή η συνεργασία, η δικαστική, θα ε, συνεχιστεί γιατί δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά αυτά που είναι στον Ειδικό Ωκεανό. Αυτό θέλω να το ρωτήσω εγώ, αλλά τώρα δεν με τι συνάδελφοι θέλω να σα ρωτήσουν. Κύριο Γκέλλερ πρώτα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Ποπόφσκι. Ελπίζουμε όλοι ότι με τον σχεδιασμό σας στο μέλλον θα φτιάξετε ένα οργανόγραμμα που θα είναι πλήρες, δεν θα υπάρχει λέξη vacant πλέον, άδεια θέση, θα είναι όλες οι θέσεις κατηλημένες γιατί οι κρίσεις δεν μας περιμένουν πέφτουν επάνω μας ε, και ελπίζω να μην σχεδιάζεται κάποια επανάσταση, αλλά ελπίζω να σχεδιάζεται πώς θα αντιδράσουμε στις επαναστάσεις ε, στις γειτονικέ μας περιοχές. Θέλουμε η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πολύ συγκεκριμένη και η άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν απάντησε κατά την άποψή μου σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν. Τι μπορεί ο κύριος Γιώτσο να ήθελε να εννοεί με τα ε, στρατιωτικά μέτρα είναι κάτι ενδιαφέρον. Είναι ξεκάθαρο ότι μια χώρα όπως η Λιβύη στο τέλος της επιδοχής Καντάφη γίνεται ένα failed state. Ε, είδαμε την κατάσταση στην Τινεσία. Ίσως ε, να έχουμε και στην Αλγερία κάτι αντίστοιχο, όπου έχουμε το state hook. Ε, ο Καντάφη είχε μια συνοχή στη δικαιολογία μετά από αυτό έχουμε το δυναμικό για ένα failed state. Και φυσικά υπάρχουν και χιλιάδες αυτοί μετανάστες που είναι στο δρόμο προς το βορρά, κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε για το συμφέρον των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, γιατί είναι στην γειτονιά μας όλα αυτά. Τα Ηνωμένα Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να κάνουν αυτά που, χρειάζονται, που χρειάζεται να γίνουν. Υπάρχει ανθρωπιστική διάσταση, αυτό πρέπει να γίνει βραχυπρόθεσμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέσω του Ερυθρού Σταυρού ή του Ισερυθρής Μισελίνου, στην την Εσία, στην περιοχή. Τι γίνεται όταν περνάει ο κόσμος από τα σύνορα, λίγο πολύ μένουν μόνοι τους γιατί δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν τέτοια πράγματα να τα σχεδιάσουμε. Ελπίζω ότι, ότι το Ευρωπαϊκό στρατιωτικό επιτελείο θα έχει κάποιο σχεδιασμό και για ανεπιθύμητες εξελίξεις. Δηλαδή τι κάνουμε αν τελικά εκτελέσουν τον Καντάφη οι πολίτες του. Τι κάνουμε αν ε, πάρουν ε, ομήρους Ευρωπαίους, όπως είχε γίνει με τον Σαντάμ Χωσέιν. Υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις και πρέπει να τα σχεδιάσουμε όλα αυτά, να έχουμε στο μυαλό μας ένα πλάνο. στην, για τη δυνατότητα συντονισμού, λοιπόν, θα ήλπιζα ότι όλοι οι πολίτες από τα 27 κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να είναι ασφαλείς Όλοι, όλα τα κράτη-μέλη έχουν πολίτες εκεί, κάποιοι έχουν στείλει πλοία και αεροπλάνα ενδεχομένω. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκολτιέρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Ποπόφσκι. Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι η πρώτη μια μακρά σειρά συναντήσεων, δεδομένων και των αρμοδιοτήτων που έχετε εσείς στην υπηρεσία. Είστε ουσιαστικά ο συνδιαλεγόμενος ε, φύση και θέση αυτής της ε, Επιτροπής. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη Λιβύη και να φτάσω στο θέμα της οργάνωσης υπηρεσίας και δεδομένης της ε, κατάστασης και των συγκεκριμένων προβλημάτων που υπάρχουν. Μου φαίνεται ότι το όλο θέμα της Λιβύης, βέβαια όλο αυτό θα το μπορούσαμε να το διευρύνουμε για όλη τη Βόρεια Αφρική, είναι ένα πρακτικό παράδειγμα αυτό που δεν έχουμε και αυτό που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι οι πληροφορίες. Διαβάζοντας λίγο προσεκτικά τον τύπο, δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, υπάρχουν κάποιες φωνές ε, και υπάρχει μία ε, αλληλοεπικάλυψη και δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα. Δεν ξέρω κατά πόσον ε, η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει κάποιε πιο αξιόπιστες πληροφορίε για τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη. Αυτό σα το λέω διότι υπάρχουν ε, διάφορες εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Είναι σαφές ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε υπέρ της δημοκρατικής εξέλιξης της κατάστασης, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τη δολοφονία ανθρώπων, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ε, δημοκρατική ε, πορεία της Λιβύης και του λαού της. Το να γνωρίζουμε αν συνέβησαν ή αν είναι εξελίξει βομβαρδισμοί πολιτών ε, μέσω αεροσκαφών, είναι σημαντική είδηση, διότι ε, συζητείται το κατά πόσον θα έχουμε μια no-fly zone. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν συνέβησαν πράγματι ή όχι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αν τα θύματα είναι 300.000 ε, τα οποία αναφέρουν κάποιες οργανώσει ή πάνω από 10.000 ε, που αναφέρουν κάποιε άλλε πηγέ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιε οι διαφορές, οπότε πρέπει να έχουμε κάποιε πιο αξιόπιστε πληροφορίε για να δούμε ποιο είναι ο πολιτικός μας προσανατολισμός, να καταλάβουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Και δίνεται η αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν είναι και πολύ καλά εξοπλισμένη ε, για την κατάσταση αυτή. Εμείς δεν ξέρουμε πόσα θύματα υπήρξαν και δεν ξέρουμε και τι απάντηση υπήρχε ή είναι εξελίξη ε, και τι ε, έγινε κατά των διαδηλωτών. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στην κατάσταση της Λιβύη, ε, λόγω της ιστορίας, ε, των φυλών. Είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά για τη Λιβύη και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε περαιτέρω προσοχή, διότι εμείς χρειαζόμαστε τα πάντα εκτός από μια νέα Σομαλία η οποία θα βρίσκεται και στο Μεσόγειο. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο φαίνεται ότι δεν διαθέτουμε είναι η οργάνωση. Καταρχάς μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, ένα ε, κράτος το οποίο είναι επικεφαλής. Δεν υπάρχει αντιπροσωπεία, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος ο οποίος ε, να αναλάβει τα ενία. Πώς μπορούμε να λέμε ας επαναπατρίσουμε τους πολίτες. Θα ήθελα να ξέρω τι ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχουν εθνικές ανεξάρτητες δράσεις οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ των επαναπατρισμού πολιτών διότι δεν υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα αναλάβει τον οργανωτικό ρόλο επιτόπου. Θα υπάρξει λοιπόν ε, ένα κράτος το οποίο θα αναλάβει ως επικεφαλής ή όχι στη Λιβύη. Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουμε και τι δομές ε, υπάρχουν. Είπαμε τι κάνει το MIC, τι κάνει το στρατιωτικό επιτελείο. Και αν αυτές οι πρώτες συνεδριάσεις αυτής της task force, ε, αυτής της ομάδας οδικών καθηκόντων στην οποία αναφερθήκατε, άπτονται αυτού του ε, Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο είναι υποσυζήτηση και το οποίο ελπίζω να γίνει και στο οποίο αναφερθήκατε στο πρώτο τμήμα της παρέμβασής σας. Διότι θα πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος συντονίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ακολουθεί την ίδια λογική με πολλούς άλλους οργανισμούς. Όλοι θέλουν να υπάρξει συντονισμός, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται ο συντονισμός. Είναι κρίμα λοιπόν που δεν διαθέτουμε τρόπου συντονισμού και δεν υπάρχουν ε, αποτελέσματα αυτή τη στιγμή συντονισμένης προσπάθειας από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με μονομένε δράσει από κράτη-μέλη. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό στο ενδεχόμενο να πάμε πέραν των όσων λέει το ψήφισμα 1970 για τον τύπο της δράσης αλλά και για μια no-fly zone, αλλά όλα θα εξαλτηθούν με, από το τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου. Δεν θα επανέλθω στα άλλα σημεία, διότι συνδέονται και με το επόμενο σημείο που έχουμε στην ημερία διάταξη. Στην έκθεσή μου αναφέρεται το επιχειρησιακό αρχηγείο και να πω κάτι τελευταίο από αυτού. Από ό,τι κατάλαβα από την απάντηση της είπα της εκπροσώπου Άστον στην πρωτοβουλία της Βαϊμάρης, υπάρχει μια καινοτομία. Αναγνωρίζεται η ανάγκη ενός επιχειρησιακού στρατηγίου, αλλά λέγεται ότι αυτή η ανάγκη θα πρέπει να αξιολογηθεί όσον αφορά το κόστος και το όφελος. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση λοιπόν αυτού του κόστου ωφέλου ε, για την ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια δομή και σε σχέση με τι πέντε υφιστάμενε δομέ και κατά πόσο θα πρέπει να ξεκινήσει μια πρακτική διαδικασία για να γίνουν όσα είπε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο ότι πρέπει να γίνουμε. Να εξετάσουμε δηλαδή το δυνατότητα να υπάρχει ένα επιχειρησιακό αρχηγείο με βάση τη σχέση κόστου ωφέλια. Monsieur le president la parole. Ευχαριστούμε, ο Λίζεκ ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα πολωνικά να σας το πω, αφού μπορώ. Παρά το ότι δεν είναι τόσο δημοσιογράφος να λέμε τη μητρική μας γλώσσα. Τέλος πάντων, έχω δύο-τρεις ερωτήσεις. η μία θεσμικού στατικού χαρακτήρα και άλλη μία πιο συγκεκριμένη ερώτηση έχω. Πρώτα πρώτα το εξή. Ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες της ε, Σύνθηκης της Λισαβόνας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θα πρέπει επίσης να σας πω κάτι για την απερχομένη ε, Πολωνική Προεδρία και την επόμενη, την Ουγγρική που ακολούθησε. Για θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής αυτό το οποίο έγινε ήταν αυτό το οποίο ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρο τη χώρα μα, ο πρωθυπουργό τη χώρα μα, μάλλον και οι παίκτε τη χώρα μα, ότι θέλουν να προωθηθεί αυτή η πολιτική, θέλουν να υπάρξουν βήματα πρόοδου. Δεν, λέω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε λεπτομέρειε για το τι γίνεται, όμω θα πρέπει να μα πείτε, αγαπητέ, εσεί και η ε, κυρία Άστον, Πώς φαντάζεστε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Προεδρία όσον αφορά την ε, πολιτική ασφάλειας και την εξωτερική πολιτική. Έχετε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά αυτή την συνεργασία. Επομένως, θέλουμε με την Ουγγρική Προεδρία που θα έχουμε την Προεδρία να ξέρουμε τι θα γίνει. Τώρα κάτι άλλο, μάλλον στρατηγικό χαρακτήρα. Σε σχέση με αυτή την σύμπραξη, τη συνεργασία μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ακούγονται πολλά, πολλές απόψεις όσον αφορά τις συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Γίνονται και διάφορε πάρα πολύ σημαντικέ ε, ανακοινώσει και δηλώσει για το ότι χρειάζεται να υπάρξει συντονισμό και συνεργασία συνεργασία στενή. Όμως εσείς για πετε μας, πώς βλέπετε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Για να δούμε επομένω. Τι αποφάσει να και σε ποιο επίπεδο συνεργασία και εσεί προσωπικά πώ θα εμπλακείτε ε, σε αυτή τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωση Έχω και μια άλλη ερώτηση, τρίτη, πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ξέρετε, είμαι ο εισηγητής κάποιας ε, έκθεσης που αφορά την Γεωργία. Τα πράγματα σχετικά σταθεροποιήθηκαν στη χώρα. Έχουμε και τη συμφωνία του 2008, η οποία όμως ακόμη δεν έχει τηρηθεί στο 100% και ξέρετε ότι οι παρατηρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στις περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι, δηλαδή στην ε, Νότιο Οσετία. Μου του την Αμπγάζη. Επομένως, για πέστε μας εσείς, από όσα ξέρετε, τι γίνεται. Ευχαριστούμε, ως Μπουτικόφερο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, ίσως δεν το κατάλαβα σωστά κύριε Παπαυσκή, αλλά η πλατφόρμα κρίσης, crisis platform που αναφέρατε, ποια σχέση θα έχει με την Επίτροπο Κρίσεων που έχουμε και κατά πόσο τελικά είναι αλλολοεπικάλυψη ή όχι. Δεύτερον, σχετικά με τις λέξεις pooling και sharing. Μέσα στα πλαίσια της ε, άτυπης συνεδρίασης έπαιξε κάποιο ρόλο. Αναφέρθηκε στη συνεδρίαση ως ε, θέμα και ήθελα να μάθω ε, ποια ήταν τα συγκεκριμένα βήματα που τελικά προβλέφτηκαν και ποια να μας τα αναλύσετε. Για την Λιβύη, το 2006 ήδη υπήρξε μια κοινή άσκηση Η VAC06 ήταν ε, το κωδικό όνομα, μέσα στα πλαίσια της οποίας κάποιες χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες ε, μπορούν να ε, εκενωθούν, να επαναπατριστούν φεύγοντας από μια χώρα της, που δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν κάποιες τέτοιες ταραχές. Λίγα χρόνια μετά βλέπουμε de facto ότι υπάρχει στο ΝΑΤΟ μια τέτοια ε, δράση. Υπάρχει μια κοινή δράση Γερμανίας ε, και Μεγάλης Βρετανίας ε, μυστική η οποία εκενώνει πολίτες και θέλω να ξέρω εφόσον πριν από πέντε χρόνια έγινε αυτή η άσκηση ποια είναι αυτά ε, που τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή στην πράξη εφαρμόστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει τις κυρώσεις ε, ΟΗΕ. Αυτό δεν το θεωρώ λάθος, αλλά όχι όμως και επαρκές. Το θέμα της no-fly zone, της ε, ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, η ύπατη εκπρόσωπος είναι υπέρ του να συζητήσουμε και την εφαρμογή κάτι τέτοιου με τους εταίρους ή όχι. Η Αμερικανική κυβέρνηση ε, ήδη προσπαθεί να το κάνει. Στη Γερμανία υπάρχουν ε, διφορούμενες απόψεις. Ε, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή της και πώς θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Καντάφη, όπως και στο παρελθόν, έχει τώρα την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει χρήματα, να πληρώσει και να φύγει, γιατί δεν υπάρχει αυτό το no-fly zone. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα το μόνο που κάνει είναι να ε, υιοθετεί τις κυρώσεις ε, του ΟΗΕ και γιατί δεν πάμε παραπέρα, πραγματικά αυτό το αναρωτιέμαι. Να υπάρχει αυτή η απαγόρευση πτήσεων και πάγωμα των ε, συναλλαγών. Για τη Σομαλία τώρα, αν κατάλαβα σωστά, υπάρχει μια τρίτη ε, επιχείρηση μετά την Αταλάντα και την UTM υπάρχει μια δεύτερη UTM για την ε, για τις περιπολίες της ακτές της Ομαλίας. Αυτό που δεν άκουσα είναι μια κριτική, μια αντιπαράθεση κριτική για το γεγονός ότι de facto τους τελευταίους μήνες όλα όσα κατάφερε η Αταλάντα ήταν να γίνει η πειρατεία ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο στη Σομαλία και όχι να σταματήσει. Είναι ένα business model επιτυχημένο αυτό στη Σομαλία σήμερα όπως ήταν και πριν από ένα χρόνο. Πραγματικά δεν πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Ε, τι γίνεται, πώς θεσπίστηκαν όλα αυτά. Στο εσωτερικό της χώρας ε, ε, υπάρχουν πολλοί που εξαρτώνται από αυτή την κεντρική βιομηχανία της πειρατείας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που είπε η κυρία Άστον ότι θέλει μια γενική στρατηγική να συζητηθεί. Ξέρει καθόλου ε, πώς θα είναι αυτή η στρατηγική, ποια μορφή θα έχει. Και το τελευταίο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε τις εξελίξεις στις αραβικές χώρες πολλές φορές άφωνοι. Ε, υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πτήσεις που κάποιοι έχουν πάρει, όμως από στρατηγική άποψη και ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη αυτού του κύματος επαναστάσεων που δεν έχει τελειώσει, αυτό δεν έχω ακούσει από κανέναν πώς θα αντιμετωπιστεί. Πρέπει πραγματικά να δούμε ε, πώς θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο και πώς θα το λύσουμε. Η κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω ένα ερώτημα σχετικά με τη Λιβύη. πόσο μακριά έχει πάει το θέμα της απαγόρευσης πτήσεων και πώς θα εφαρμοστεί. Πρέπει να γίνει στρατιωτική εφαρμογή. Και επίσης, άλλο ένα θέμα, έχει να κάνει με το στρατιωτικό στην Αιγυπτό και στην Τινησία, αν θα ε, εμπλακούν και αυτοί. Σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακριβώς θα γίνει η στρατιωτική επέμβαση. Αν δούμε πόσο εξοπλισμένη είναι αυτή η χώρα, η Λιβύη, χωρίς ε, καν τη βοήθεια των ευρωπαϊκών χωρών, να το ξαναπούμε αυτό, όπως για παράδειγμα μια απαγόρευση πτήσεων η οποία σχετίζεται με τους βομβαρδισμούς. Νομίζω ότι όλα αυτά ε, ε, οδηγούν στον κίνδυνο ενός εμφυλίου πολέμου. Αυτά τα έχουμε υποτιμήσει, νομίζω. Αυτό που πάντοτε αναρωτιόμαστε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έχουμε κάποιο θετικό παράδειγμα από το παρελθόν, αν τελικά υπήρξε μια θετική εξέλιξη ε, σε σχέση με την ε, απαγόρευση πτήσεων. και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κατάσταση η οποία δεν έχει βοηθήσει στη βελτίωση των συνθήκων ε, διαβίωσης του κόσμου. Άρα όταν μιλάμε για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να κοιτάμε λίγο και το ιστορικό, ε, πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, βήμα 1, βήμα 2, πώς θα συνεχίσει και να εξετάζουμε και τις μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις μιας παρέμβασης. Επίσης έχω ερώτηση για τον προϋπολογισμό ανθρωπίνων κρίσεων και διαχείρισης κρίσεων. Στις 10 Φεβρουαρίου οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν ότι υπάρχουν σκέψεις ή προϋπολογισμοί για τη, να, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διαχείρισης ε, κρίσεων να συγχωνευτούν. Ε, υπάρχει τέτοιο σχέδιο λοιπόν και τι πιστεύετε εσείς για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε κύριο Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εσάς κύριε Πόβος, και ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα να μας τα πείτε εδώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να ενεργήσει με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Όμω για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ε, πληροφορίε. Και όπω ξέρετε δεν έχουμε υπηρεσία πληροφοριών στην ε, Ένωση. Άρα θα ήθελα να μου πείτε αν ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ε, κρατών μελών εάν μοιράζονται τις πληροφορίες τους ε, από αυτά τα οποία ξέρουν και να μην δουλεύουμε μόνο με τα όσα μας λένε οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ. Επομένως σας ερωτώ, έχουμε κάποια συγκεκριμένα σενάρια και συγκεκριμένα πλάνα, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά ιδίως όσον αφορά την ζώνη, την επιβολή μόνο της ζώνης απογραφητήσεων και ε, όλα αυτά τα οποία αναφέραμε για τους πυράβλους, τι γίνεται. Είναι δυνατόν να, να, να, να έχουμε ευαισθησία, είναι δυνατόν να είμαστε τρωτοί όσον αφορά την επικράτειά μας να μην μπορούν να χτυπήσουν. Επομένω, για πέστε μας, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τους πυράβλους, τι θα κάνει. Και ε, βεβαίως, το θέμα δεν είναι μόνο κατά πόσο μπορούμε να αντιδράσουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων ε, κάποιο είδου ε, πληροφορίε για να έχουμε κάποιο είδου ε, πλάνα να έχουμε κάποια σενάρια προγραμματισμένα. Επομένως, για πετε μας, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες επαφές με την ε, ας πούμε προσωρινή κυβέρνηση, προσωρινές αρχές, πώς με αυτούς τέλος πάντων που, που κάνουν κομμάτι στην Δεγκάζ, δεν ξέρω πώς να τους αποκαλέσω. Τι γίνεται, έχουν ζητήσει κάποια βοήθεια, ε, μπάστε και θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποια αποστολή ανθρωπιστική, στρατιωτική στη Λιβύη. Μια που από πλευρά εκείνων των ανθρώπων ε, που κάνουν και κουμάντο στη Βεγγάζη έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Ναι. Κύριε μου το λόγο. Έχω κάποιε ερωτησούλε. Όσον αφορά την αποστολή στη Σομαλία, τι έγινε με αυτούς τους στρατιώτες. Πρόκειται για 900 που το έχουν εκπαιδευτεί. Τι έγινε με αυτούς. Επίσης όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων που αναφέρατε για το σχετικό όργανο Τι θα γίνει σε περίπτωση κάποιες κρίσεις. Ναι, όντως χρειάζεται κάποια δομή πάγια. Ένα σώμα διαρκούς λειτουργίας. Δηλαδή, συνέχεια λειτουργεί και όχι όταν πια η κρίση φτάσει στο κατακόρυφο. Τι γίνεται τώρα όσον αφορά τη στρατηγική μας. Γκάνους έχει φύγει. Συζητούμε ήδη με τους Σύρους προσπαθούμε να επανακαθίσουμε τη σχέση μας και λέχθη πριν από λίγο καιρό ότι όλα πάνε πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω. Ο Υπουργός τρίγων της Λιβύης βρισκόταν στις Βρυξέλλες και διαπραγματευόταν αυτά τα 50 εκατομμύρια αυτή την αρρωγή για τη συνοριακή εποπτεία. Τι φύλαξε των συνόρων, τι έγινε. Μα είναι δυνατόν η χώρα να βρίσκεται στι φλόγε να, έχει ξεκινήσει και η Πανάθη και εμεί να συνεχίζουμε την ίδια ρότα. Όλα αυτά προβλέπονται για χώρε που είναι σε άλλη φυσιολογική φάση. Έχουμε στατική για Εμένη, Μπαχρέιν, Λίβανο, Συρία. Τι γίνεται. Πέστε μας. Έχετε δεν έχετε. Και αν μην έχετε πέστε μας. Τέλος πάντων κάπου, να καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχουμε όλες αυτές τις απαντήσεις, αυτές τις ερωτήσεις. Και έλα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες σας. Κύριε, από το διαγράμματος. έχετε πώς θα μπορέσετε να συγκροτήσετε αυτό το σύστημα αντιμετώπισης των κρίσεων. Μας είπατε ότι ακόμα υπάρχει προβληματισμός. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η κρίση χτυπάει ξαφνικά, δεν κάθεται να προβληματιστεί σιγά σιγά. Πάντα εξαπίνεις, συλλαμβάνει κάποιον. Είδατε τώρα τι έγινε με τις ε, παραστάσεις αραβικές χώρες. Επομένως, γίνεται να έχουμε κάποιο είδους δυναμική, ενεργητική, αποτρεπτική, αν θέλετε, στρατηγική για όλα αυτά. Τώρα όσον αφορά τη συνάντηση της Βουδαπέστης. Πρόκειται περί, περιπτώσεως αντιδράσεως που έγινε από πλευρά μας, αλλά όχι συντονισμένα. Επομένως, το ερώτημά μου είναι, έχετε κάτσε να σκεφτείτε τα σενάρια που μπορούμε να έχουμε, αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τον Λίβιο δικτάτορα ή επίσης αν, αν, αν διαλυθεί σαν κράτος, αν κατρέψουν οι θεσμοί στη Λιβύη, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για κάποιο είδους αποστολή πολιτών μεν εκεί, αλλά υποστηριζόμενοι αποστολικού, γιατί μόνοι του οι πολίτε δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά σε μια τέτοια κατάσταση. Επίση, εν κατακλείδη, αυτό που είπε ο κ. Κουαλτιέρη, προ υπογράφω, και με γιατί μα ανέφερε ότι χρειαζόμαστε Κάποιου είδου ολοκληρωμένη προσέγγιση, σφαιρική, όσον αφορά αυτή την ΚΕΠΑ. Όμως, δεν έχουμε ακόμα δείγματα ότι τέτοια πολιτική έχει αναδυθεί. Αν θέλετε, μου απαντάτε. Merci, Monsieur Popovski, avec cet ambitieux agenda. C'est vraiment très ambitieux. Je euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλα προετοιμασμένο για να απαντήσω σε όλε σα τι ερωτήσει, αλλά θα προσπαθήσω όπω και να έχει. Ξεκινώντας με την Αταλάντη και το θέμα της δικαστικής συνεργασίας, η έκθεση κ. Λάντ είναι σχετικά καινούργια και στο τραπέζι. Πολλοί υπουργοί στη Βουταπέστη αντέδρασαν με θετικό τρόπο. Αυτό που προτιθέμεθα να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε τη δυνατό την ανοικεδόμηση διανοτήτων στη χώρα. Ίσως όχι να φτιάξουμε δικαστήρια και φυλακές, γιατί κάπως θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε αυτά, αλλά έχουμε τις ε, συμφωνίες Συνεργασίες με τις χώρες αυτές, οι οποίες ε, θα ήταν και ε, χωρίς μια τέτοια ε, συνεργασία. Τώρα επίσης να πω ότι αναθεωρούμε τη θητεία της επιχείρησης, να δούμε κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επιπτώσεις αυτής της επιχείρησης είναι ε, διαρκείς. Επίσης υπάρχει το θέμα της προσέγγισης μας στην όλη περιφέρεια, στο κέρας της Αφρικής δηλαδή. Όλα αυτά είναι στην ημερησία διάταξη. Αυτή τη στιγμή ε, προετοιμάζουμε συζήτηση των Υπουργών τον ε, ε, Μάρτη, στο PSC, ΕΠΑ δηλαδή. Υπάρχει μια στρατιωτική επιτροπή. Ο κύριος Καν επίσης έθεσε πολλά ερωτήματα Αυτή η ερώτηση, αυτό το ερώτημα έχει εδώ και εβδομάδες τεθεί. Τώρα ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα. Θα δούμε λίγο και το ημερολόγιο, να δούμε πώς θα είναι έτσι οι δομές, έτσι ώστε να έχουμε δύο στάδια. Πρώτον, να σταθεροποιηθεί το σύστημα, να γίνει η στελέχωση, να εκτελεστεί και μετά τα αποτελέσματα της συζήτησης για το comprehensive approach να μας δείξουν αν χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα, αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν ακόμα. Όλα αυτά θα διαρκέσουν λίγο. Αλλά απλώς να σας πω ότι δεν καθόμαστε άπραγοι και περιμένουμε τα γεγονότα να μας ε, ξεπεράσουν και την κρίση να μας ε, ξεπεράσει. Πολλοί από εσά ρώτησαν για την πολιτική μας σε όλη την αραβική περιοχή της Αφρικής, στη Βόρεια Αφρική. Να τα πω λοιπόν όλα μαζί. Έχει να κάνει με την επερχόμενη αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Είναι κάτι το οποίο ήδη σχεδιάζαμε, αλλά τώρα έχει γίνει επίγον. Όσον αφορά στην ύπατη εκπρόσωπο, αυτό που θέλει να κάνει είναι μια πολιτική συζήτηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών στις 11-12 Μαρτίου ε, όπου θα γίνει η πολιτική γειτονία στο κεντρικό θέμα. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική και την Αγγής Ανατολή. Μετά, διμερώς, ε, ε, όσον αφορά στα κράτη, θα προσπαθήσουμε περιφερειακά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι κάτι που συζητείται. Τώρα, για συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τη Λιβύη, ε, για τα ερωτήματα που θέσατε, υπάρχει αυτή, αυτό το upgrade της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Λιβύη, η αναβάθμιση όπως θα τη λέγαμε, την οποία την έχουμε συζητήσει αλλά δεν προχώρησε. Γίνεται λοιπόν τώρα μια εξέταση, μια αναθεώρηση και αυτό που παίρνουμε ως πληροφορία από τους εταίρους μας ε, στην ε, περιοχή είναι ε, πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Έχει να κάνει και με την πολιτική συζήτηση που γίνεται τώρα για το θέμα αυτό. Ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί ερώτησαν και γι' αυτό. Τα, θέμα, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι εθνικά, δηλαδή τα αεροπλάνα, τα πλοία που θα επιχειρήσουν είναι εθνικά. Δεν μπορούμε λοιπόν ελεύθερα να αποφασίσουμε. Δεν ε, είναι, τα κρα... είναι κάτι που τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν. Εμείς μόνο μπορούμε να συντονίσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα δούμε λοιπόν πώς αυτό θα γίνει στο στρατιωτικό επιτελείο. Υπάρχει ένας τέτοιος ε, ε, κλάδος συντονισμού. Πρέπει απλώς να ενεργοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε λοιπόν πέρα από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο που κάναμε επιπρόσθετα είναι ένας, αξιωμα... ένας liaison officer, ο οποίος υπάρχει στο κέντρο συντονισμού στη Μάλτα. Ε, πρόκειται για έναν ε, σύνδεσμο, αξιωματικό σύνδεσμο του, του στρατιωτικού επιτελείου, ο οποίος ε, συντονίζει αυτές τις δράσεις επαναπατρισμού. κοιτάω λίγο τις σημειώσεις μου. Για τη Λιβύη, όπως σας είπα, είναι θέμα περιφερειακό, θα έλεγα. Έχει να κάνει με την προσέγγιση μας ε, στην περιφέρεια της Βορείου Αφρικής. Χρειαζόμαστε φυσικά περισσότερες πληροφορίες. Πολλοί κάνατε αυτή την ερώτηση. Η ανταλλαγή πληροφοριών βέβαια έχει τα όρια της. Δεν έχουμε κάποιες μυστικές υπηρεσίες και ούτε θα έχουμε. Ε, στο μέλλον, το άμεσο μέλλον. Θυμάμαι τι είχε γίνει τότε μετά τις, ε, τους στη Μαδρίτη. Είχαμε πρόσβαση, έχουμε πρόσβαση σε εθνικές πληροφορίες των κρατών μελών, ε, οι οποίοι μπορούν να μας πούν ποια είναι τα κατάλληλα μέρη που μπορεί να γίνει η κάθε δράση. Έχουν δηλαδή μία πληροφόρηση από τη χώρα, αλλά πάντοτε κοιτάμε ποιος δίνει την πληροφορία. Τώρα για την ε, Λιβύη, ε, επειδή ε, δεν έχουμε αντιπροσωπεία, έχουμε μια αντιπροσωπεία στην Τίνιδα η οποία ασχολείται με τα θέματα της Λιβύης. Επιτόπου λοιπόν έχουμε συναδέλφους της ΕΚΟ που βοηθούν στις ανθρωπιστικές προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε τακτικό προσωπικό της Επιτροπής. Και έτσι λοιπόν δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά. Απλώ ε, σε συνεργασία με την Τρίπολη προσπαθούμε να έχουμε ένα συντονισμό ε, με τις πρεσβείες. Ε, βέβαια δεν έχουν όλες όλο τους το προσωπικό γιατί κάποιες χώρες το έχουν ανακαλέσει ε, κοιτάμε λοιπόν ποιοι είναι επιτόπου ε, παρόντες για να μας βοηθήσουν. Προσπαθώ να ομοδοποιήσω λίγο τις απαντήσεις για να είμαι πιο συνεκτικός στις απαντήσεις μου. Ε, οι ερωτήσεις για την ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συζήτηση, γιατί αυτό θα πετούσε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε ήδη δει ποια είναι οι αποφάσεις του, τις εφαρμόζουμε και μέσα στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούμε να πάμε παραπέρα στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων για παράδειγμα. Θα δείτε ότι υπάρχει διαφορά ε, στις, στους καταλόγους του ψηφίσματος ε, του ΟΗΕ. τη μία είναι η απαγόρευση θεωρήσεων και από την άλλη το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων που είναι πιο μικρή η λίστα. Αυτό είναι ε, μια συζήτηση που συνεχώς ε, τρέχει στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω τώρα σε ποια φάση είμαστε προς το παρόν. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση για μια συμβολή σε μια ζώνη του πτήσεων. Βέβαια, δεν χρησιμοποιούμε κανένα άλλο στρατιωτικό μέσο πέραν των αεροπλάνων και πλοίων ε, που είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να επαναπατρίσουμε τους πολίτες μας, όπως ξέρετε. Για το θέμα του των στρατιωτικών ε, και των ε, περιφερειακών ε, θαλάσσιων δυνατοτήτων. Ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τις ακτοφυλακές των χωρών εκεί, αλλά αυτό φυσικά απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τα αγράτη μελη που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και το προσωπικό, αλλά και να βρούμε και τη σωστή χρηματοδότηση. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν για παράδειγμα, είχαμε μια αποστολή κατάρτιση στη Μολδαβία, εκπαιδευτική αποστολή, η οποία ε, πέτυχε όσον αφορά ε, στην στην οικοδόμηση δυνατοτήτων ε, στην περιοχή μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας στα σύνορα. Για τα συστημικά ζητήματα τώρα που τέθηκαν από κάποιους από εσά. Πρώτον, το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού, του επιχειρησιακού στρατηγίου δεν είναι κάτι καινούριο. Το σχόλιο που έκανε ο κύριος Κουλτιέρη είναι Όντω έτσι, χρειαζόμαστε μία ανάλυση κόστους ωφέλους. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από το απλό ερώτημα του τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε να κάνουμε ώστε να είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να ε, επιχειρήσουμε σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το SHAPE, τα κεντρικά του ΝΑΤΟ, μετά έχουμε κάποια άλλα ε, αρχηγεία τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι χρειαζόμαστε, αν θα πάμε πιο πέρα. Δεν χρειαζόμαστε μια άλλη ιδεολογική συζήτηση για το ευρωπαϊκό στρατηγείο. Είναι κάτι λοιπόν που χρειάζεται να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Και τώρα θα γυρίσω στα πολωνικά για να είμαι δίκαιος. Κύριε Αντιπρόεδρε, απάντηση στα ερωτήματά σας. Καταρχάς και το ρόλο της κυλιόμενης ε, προεδρίας είναι σχετικά περιορισμένος. Είναι μεν. Είπατε εκπρόσωπος ε, που ε, θέτει τις προτεραιότητες και αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με την κυλιόμενη προεδρία, το προεδρεύονται κάθε φορά. Αυτό που κάνει η κυρία Άστον είναι να συζητά πάντοτε, ώστε να βρίσκονται τα σημεία ενδιαφέροντος που αφορούν σε κάθε κράτος μέλος. Τι είναι αυτό που ενδιαφέρει το κάθε κράτος μέλος. Όμως πάντοτε συζητούμε πολλές φορές μέχρι να μπει κάτι στην ημερήσια διάταξη, γιατί η ημερήσια διάταξη είναι δική μας, είναι αυτή που θεσπίζεται από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κάπως έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει και στο μέλλον λοιπόν και χαιρόμαστε που η Πολωνική Προεδρία θεωρεί το θέμα της ε, ασφάλειας και της άμυνας ως προτεραιότητα γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά θεμάτων. Όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ, εγώ γνωρίζω προσωπικά τους περιορισμούς που υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν πως μπορούμε να συζητήσουμε σε επίσημο επίπεδο, να συζητήσουν τα δύο όργανα μεταξύ τους, να γίνει δηλαδή μια ανταλλαγή απόψεων και είμαι πολύ ανοιχτός ως προς το να ενημερώσω τους ε, πρέπει του ΙΣΕΠΑ και τώρα για την αποστολή στη Γεωργία είναι μια χρήσιμη αποστολή, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που μπορεί να έχει, γιατί είναι η μόνη αποστολή στην περιφέρεια αυτή. Βέβαια έχουμε πρόβλημα πρόσβασης στις κατεχόμενες περιοχές και υπάρχουν και τα μέρη που συνδιαλέγονται στην, ε, στη Γενέβη υπό τον Πιέρ Μοντέλ, τον ειδικό μας εκπρόσωπο Πρόκειται για ένα φόρουμ όπου ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όμως, ε, όπως και να έχει, η αποστολή στη Γεωργία είναι, είναι ενδράση και είναι και η μόνη αποστολή της Ευρωπαϊκής ε, ε, διεθνής μάλλον παρουσία στην περιοχή. Τώρα για τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εμείς έχουμε το δικό μας κομμάτι. Είμαστε και της κυρίας Γεωργίευα. Είμαστε εμείς αυτοί που κάνουμε το δικό μας κομμάτι και μαζί με την Κομισιόν συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να συνδυάσουμε διάφορα ε, οργαλεία που έχουμε όπως αυτό το Crisis Coordination Shell στο Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο. Απ' την άλλη έχουμε τη Γενική ε, Διεύθυνση ΕΚΟ και το εργαλείο ΜΙΚ, τα οποία τα έχουμε και λαμβάνουν χώρα, για το pooling και το sharing. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχουν ε, λεπτομέρειες που να γνωρίζω για να σας δώσω. Έχουμε συζητήσει με τους αρχηγούς επιτελείου, τους γενικούς επιθεωρητές ή τέλος πάντων όπως ονομάζεται σε κάθε χώρα Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ε, δυνατότητα και όταν στο τέλος την ορίσουμε, στα τέλη Μαΐου ελπίζουμε με τους Υπουργούς Άμυνες να έχουμε ένα πιο ε, πλήρες ε, τοπίο θα έλεγα. Για την ακτοφυλακή για την ε, φύλαξη των ακτών στη Σομαλία και την ε, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων έχω ήδη μιλήσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει πρώτα να επιτευχθεί κάποια πρόοδο για αυτά που έχουμε για να σταθεροποιήσουμε τις δομές μας και κατόπιν να το αναπτύξουμε περαιτέρω, ανάλογα με την κατάσταση. Όσον αφορά τώρα την ολοκληρωμένη προσέγγιση, αυτή είναι σαφώς μια μεγάλη πρόκληση. Προς το παρόν, εμείς είμαστε παρόντες με τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά πλέον όλα τα μέσα είναι ομαδοποιημένα σε ένα σημείο στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, και η άμυνα και η ασφάλεια και η ανάπτυξη παρεπιπτόντως, διότι έχουμε και μια κάποια ευθύνη για τον προγραμματισμό της αναπτυξιακής βοήθειας που, θα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάπτυξη ε, αντιμετώπισης κρίσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Γκουαλτιέρη, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, Μία παρατήρηση μόνον, διότι εγώ είχα κάνει μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το θέμα των θυμάτων και τη χρήση βομβαρδιστικών αεροσκαφών ε, για βομβαρδισμούς πολιτών στη Λιβύη. Το γεγονός ότι δεν μου απαντήσατε σημαίνει ότι δεν έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες επί του θέματος ή ότι αυτές οι πληροφορίες είναι διαβαθμισμένες, επομένως ε, δεν μπορείτε να μας δώσετε τις πληροφορίες γιατί δεν είναι και κλεισμένο των θυρών η συνεδρίαση. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Έχουμε κάποιες εκτιμήσεις. Βασιζόμαστε στις πληροφορίες ε, που λαμβάνουμε από τους δορυφόρους Ίτσεν και από τα κράτη-μέλη. Και έχουμε και επίσημα εντό εισαγωγικών ε, στοιχεία από πλευρά Λιβύης. Τα επίσημα στοιχεία, αν μπορούν να είναι επίσημα, είναι 300 άτομα. Αλλά έχουμε και στοιχεία τα οποία βασίζονται σε πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται επί τόπου και μας λένε ότι ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 600 και 3.000 αλλά και πάλι είναι πολύ δύσκολο να επαληθεύσουμε αυτά τα στοιχεία, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αξιόπιστα. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε ότι θα πρόκειται και την πρώτη από μια σειρά από επαφές και συζητήσεις μαζί σας για να μπορείτε να μας ε, ενημερώσετε όσον αφορά το τι γίνεται με την εξωτερική δράση για όλες τις επιμέρους επιχειρήσεις. Όχι δεν θα συζητήσουμε άλλο γιατί ήδη ε, τα είπαμε με αρκετή πληρότητα. Καλά τέλος πάντων. Θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό. Πραγματικά όμως ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σφανόρντε. Τι λέει ο κύριος αναπληρωτής. Όσον αφορά αυτή τη δαπάνη των 10 εκατομμυρίων που γίνεται από την υπηρεσία του για εξωτερικές, για, συγγνώμη, για δημόσιες σχέσεις γιατί είχε ανυποσχεθεί ότι τελικά θα πρόκειται για μια δράση ουδέτερη δημοσιονομικά. Όχι, δεν έχω λεπτομέρειες, τι να σας πω. Τώρα ξεκινήσαμε τη λειτουργία αυτής της ομάδας επικοινωνίας και όταν λέω ομάδας δεν θα είναι και τόσο μεγάλη. Θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε. Θέλουμε ποιο μας να λειτουργεί καλά. Αυτά είναι τα μέσα σχέδια μας, αλλά όχι δεν θα είναι τόσο ψηλή δαπανή όσο είπατε. Κύριε Έχω μία ερώτηση. κύριε Έχουμε διάφορα στρατηγία όπως είπε αλλά είναι όλα του ΝΑΤΟ. αν χρειαστεί να αναλυθεί δράση για να υποστηριχθεί για κάποιο είδου πολιτική επανέμβαση, τι θα πρέπει να γίνουμε. Όχι, αυτό δεν το έχουμε ήδη προγραμματίσει. Εάν γίνει κάτι, θα είναι το στο πλευρά του ΣΕΠ, θα είναι στρατιωτική επιχείρηση. Για τη στρατιωτική επιχείρηση, μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε το ΣΕΠ, αλλά Άρα αναπερίπτωση θα αποφασίζουμε για το ποια βάση, ας το πούμε, ποιες καταστάσεις θα χρησιμοποιήσουμε. Πότσλαμ, Παρίσι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Και έχουμε και άλλα στρατηγικά, και, άλλα στρατηγικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εξαρτάται από το κράτος μέλος, πρόεδρος. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, nous reprenons euh, les travaux avec euh, le rapport de monsieur. Παρακαλώ, συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Κουαλτιέρη για την ε, εξέλιξη της πολιτικής ε, ε, κοινής ασφάλειας και άμυνας. Υπήρξε μια καθυστέρηση στη μετάφραση, όμως τώρα είναι διαθέσιμη η έκθεση. Σας θυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Κατάθεση τροπολογιών 8 Μαρτίου, επόμενη εβδομάδα. Και στις 15 Μαρτίου τελευταία εξέταση, οπότε στις 12 Απριλίου θα γίνει και η ψήφιση στην Ολομέλεια, αλλά κύριε Κολθίρη, έχετε... Στην Επιτροπή Εξωτερικών, συγγνώμη. Είχε γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον φλεβάρι. Ελπίζω ότι σας ε, δώσαμε στοιχεία σχετικά με τα συγκεκριμένα σημεία της έκθεση και όχι με τις φιλοσοφικές απόψει του καθενός. Ε, γνωρίζουμε τις θέσει του καθενός. Να πάμε λοιπόν κατευθείαν στο ψητό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα κάνω μία εισαγωγή, μια σύνοψη εν είδη εισαγωγής, ε, διότι υπάρχει πλέον ε, η έκθεση, ε, επομένω δεν χρειάζεται εγώ να την αναφέρω αναλυτικά. Να σας πω απλώς ότι υπάρχουν κάποια μικρά σημεία στα οποία η αγγλική μετάφραση χρήζει παρεμβάσεων, διότι υπάρχουν κάποιες εκφράσεις οι οποίες είναι λίγο πολύ λέξη μετάφραση και δεν ε, εκφράζουν ακριβώς αυτό το οποίο εννοούσα. Ζητώ συγγνώμη αν υπάρχουν ατέλειες λοιπόν. Ε, φιλοδοξώ να διορθωθούν. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία επί τούτου δεν έχω συμπεριλάβει στην έκθεση και φυσικά κάθε συνάδελφος έχει δικαίωμα να προτείνει να συμπεριληφθούν ε, κάποια στοιχεία εν είδη τροπολογιών. Δεν έχω αναφερθεί σε επιτυχίες και λόγω του γεγονότος ότι είναι αρκετά μακροσκελής η έκθεση που αφορούν κυρίως ε, εξωτερικά σενάρια παγκόσμιας ασφάλειας αντιπυραυλική άμυνα, η απειλή από το Ιράν, θέματα στα οποία ήδη έχει εκφράσει την άποψή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφέστατα και επομένως δεν έχω επαναλάβει στοιχεία τα οποία δεν θα είχαν ε, προσδώσει κάτι το νέο, αλλά επικεντρώθηκα απλώς και μόνο στο θέμα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μετά τη συνθήκη της και επειδή η ουσία της έκθεσης, ε, όπως θα διαπιστώσατε ελπίζω, είναι ότι υπάρχει ανάγκη μιας πιο ισχυρής ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα συνδέει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την ε, ΚΕΠΑ και τις υπόλοιπες πτυχές ε, της εξωτερικής δράσης. Γι' αυτό ακριβώς εσκεμένα παρέλειψα μια ανάλυση εξωτερικής πολιτικής των διαφόρων θεάτρων επιχειρήσεων, θεωρούσα, θεωρώντας ότι ε, αυτό, θα έπρεπε να αναφέρεται στην έκθεση κοινή εξωτερικής πολιτικής και όχι της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τώρα, επειδή υπάρχουν εξελίξεις στις χώρες από την άλλη πλευρά της Μεσογείου, των βορειοαφρικανικών χωρών, τη Λιβύης που συζητήθηκαν, ίσως ε, μέσω τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν ε, υπήρχαν αρχικό στο κείμενο. Πέραν αυτού, eh, Λοιπόν, η έκθεση συνδέει την εξέλιξη των προκλήσεων που θέτει το Διεθνές Σύστημα στην ασφάλεια, που πρόκειται για νέες προκλήσεις και αφορούν νέες πτυχές της ασφάλειας, με τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Συνδέονται λοιπόν αυτές οι δύο πτυχές και συνεπώς αναφέρεται η ανάγκη να γίνει ένα τεράστιο άλμα για να υπάρχει μια αποτελεσματική ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα ασφαλείας. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα θεωρεί ότι η ασφάλεια είναι εγκάρσιος στόχος ε, στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεωρεί ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι μέσο αυτής της πολιτικής. Προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο οι διάφορες θεσμικές, πολιτικές, οργανωτικές ε, και άλλα πτυχές πρέπει να το μετωπιστούν ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να κάνει αυτό το άλμα. Διότι η συγκεκριμένη προσέγγιση προς το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι μια ξεχωριστή τομεακή πολιτική αλλά και να τη συμπεριλάβουμε πλέον σε μια πλήρη δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και από πλευράς για τον τρόπο προς τον οποίο συνδέομαι τα διάφορα όργανα και υπηρεσίες, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο ε, συνδέουμε διαφορετικές ε, νομικές βάσεις και διάφορα ε, νομικά μέσα που αφορούν το κοινοτικό πλαίσιο και το συγκεκριμένο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και της ΚΕΠΑ και τις σχέσεις μεταξύ ευρωπαϊκής διάστασης και κρατών μελών. Πρόκειται για μια περίπλοκη προσπάθεια και Επ' αυτού αναπτύσσει κάποιες σκέψεις η έκθεση. Υπάρχει η πρόταση λοιπόν να προχωρήσουμε περαιτέρω και να συνδέσουμε με την Ευρωπαϊκή Πολιτική ε, Ασφάλειας και Άμυνας και μία στρατηγική στη βάση ενός ε, πολιτικού πλαισίου και στρέφομαι προς τα κράτη-μέλη για να δούμε τι έγινε στον πρώην τρίτο πυλώνο των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης με τη διαδικασία που ξεκίνησε μέσω της συνθήκης του Σέγγεν και μας βοήθησε στο να έχουμε ε, πραγματικές... Ε, προσπάθειες από πλευρά κρατών μελών και τώρα έχουμε κάτι αντίστοιχο με την ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας και υπάρχει και άλλη πτυχή που αφορά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και η υποεπιτροπή μας θα πρέπει να ζητήσουμε και για τον άξονα της ασφάλειας και της άμυνας. Η άλλη πτυχή τώρα είναι το θέμα της εμπλοκής και της δυνατότητές μας να διαδραματίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πολιτικό ρόλο. Διότι όταν μια πολιτική ασφάλειας ε, περιλαμβάνει και άλλες πτυχές και πάει πέραν ε, των πτυχών της εξωτερικής ε, δράσης, θα πρέπει να συνδυάσουμε την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πτυχή της ΚΕΠΑ, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτελεσματικό αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει τεράστια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί αλλά και θα πρέπει να διαδραματίσει ένα πιο ε, σημαντικό ρόλο από την ε, ανάγνωση κατά γράμμα του άρθρου 36 της Συνθήκης της Λισαβόνας και επειδή έχει και ρόλο νομοθέτη θα μπορεί στη συνέχεια να δει και την εφαρμογή μιας αποφασιστικής πτυχής της ευρωπαϊκής δράσης, η οποία θα έχει επιπτώσεις ε, ε, σε όλες τις πολιτικές ασφαλείας από πολλές πτυχές. Θα πρέπει να υπάρχει και μια στενή συνεργασία της υποεπιτροπής μας με άλλες επιτροπές ε, που άπτονται πολύ σημαντικών πτυχών της ασφάλειας, κυρίως της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά και της Επιτροπής Ήτρε, για παράδειγμα. Κατόπιν υπάρχει ο ρόλος της είπα της εκπροσώπου, η δυνατότητα να υπάρχει μια στενα, πιο στεναρή σχέση και να δημιουργηθεί μια πολιτική συνένεση, εκμεταλλευόμενη και πλήρως τις δυνατότητες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, να υπάρχει πλήρη εμπλοκή των οργανισμών της και των προσωπικότητων της, αν θέλετε, να μπορέσουμε έτσι να προετοιμάσουμε μια πολιτική συνένεση και η ύπατη εκπρόσωπος να έχει ένα πιο ισχυρό ρόλο ε, ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και στις επαφές της με τους Υπουργούς Άμυνας. Υπάρχει και μια οργανωτική πτυχή που αφορά την οργάνωση της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εδώ ξεκίνησε ήδη η συζήτηση στο προηγούμενο ε, σημείο που είχαμε στην ημερήσια διάταξη. Στην έκθεση υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει πραγματικά αυτό το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων, που δεν θα είναι όμως ε, ένας χώρος αντίδρασης μόνο στην κρίση, αλλά θα είναι και ένα κέντρο προετοιμασίας και πρόληψης για την κρίση, προηγμένου προγραμματισμού, ώστε να τίθενται ε, γύρω από ένα τραπέζι διάφοροι παράγοντες και της υπηρεσίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεκτικοί με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της Μαδρίτης. Επομένως, μια εξωτερική υπηρεσία όχι ως ε, όργανο αλλά μια υπηρεσία στην υπηρεσία των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ε, μέσω κοινοτικών μεθόδων είτε μέσω διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει δηλαδή η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης έχει, να έχει ένα διτό ρόλο προηγμένων οργανωτικών δυνατοτήτων απάντησης στην κρίση και τη δυνατότητα να δημιουργεί ένα αμάλγαμα διαφορετικών θεμάτων και να λαμβάνονται αποφάσεις ε, μέσω μιας ε, Αλυσίδα λήψη αποφάσεων είτε με κοινοτικό τρόπο είτε δίνοντας προτεραιότητα στο Συμβούλιο ανάλογα με το ποια είναι η προεξάρχουσα φύση τη απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό όμω να βρίσκονται όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να έχουν στη διάθεσή του και κάποια ε, συνεκτικά μέσα. Δεν αρκεί μόνο ένα τραπέζι, θα πρέπει να υπάρχει ένα situation room το οποίο θα δίνει αποτελέσματα και θα υπάρχει μια δομή που θα απαντά αυτό το, γύρω από αυτό το Crisis Management ε, Board. Υπάρχουν τώρα και κάποιες πτυχές τις οποίες δεν θα σταθώ γιατί τις έχουμε επισημαίνει επανειλημμένως. Ε, η σχέση κοινή πολιτικής ασφάλειας και ε, και άμυνας, το enforcement for stability, η θέση μας και όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά τα τμήματα τα οποία θα θέλαμε να περιλαμβάνονται στην υπηρεσία. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα shared service center το οποίο θα καθορίζει με σταθερό τρόπο υποστήριξη σε πολιτικές αποστολές ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και θα μας επιτρέπει να έχουμε σταθερές δυνατότητες ως Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη δομή και τον εξοπλισμό αλλά και την ε, ε, διοικητική διαχείριση των αποστολών. Τώρα, όσον αφορά τη διάσταση της άμυνας, επισημαίνεται ότι η συνολική προσέγγιση δεν σημαίνει ότι θα πέσει σε δευτερεύοντα ρόλο η στρατιωτική πτυχή της διαχείρισης κρίσεων, που είναι ένα από τα μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Εκφράζεται μια κάποια ανησυχία ως προς το γεγονός ότι Παρά το γεγονός ότι συνήθως λέμε, συχνά λέμε ότι η οικονομική κρίση μας οδηγεί σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση του τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, ε, φοβούμαι ότι μπορεί να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Να έχουμε μείωση της ε, δέσμευσης των κρατών μελών στον τομέα αυτό, αλλά και ταυτόχρονα ελοχεύει ο κίνδυνος να μην γίνει και με συντονισμένο τρόπο. Δηλαδή, να γίνουν βήματα προ την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα επιθυμούσαμε, δηλαδή το να έχουμε καλύτερο συντονισμό και να ε, συμπεριληφθούν οι εθνικές συνεισφορές σε μια συλλογική προσπάθεια κοινή άμυνας. Δεν θα επανέλθω τώρα σε κάποιες ε, πιο συγκεκριμένες πτυχές, απλώς θα τις απαριθμίσω περιλαμβάνοντας την έκθεση το θέμα του επιχειρησιακού στρατηγίου, ε, το οποίο αναπτύσσεται λίγο περαιτέρω στην έκθεση και υπογραμμίζεται ότι αυτή η μελέτη κόστους ε, ωφελίας και το επιχείρημα που χρησιμοποίησε και η Λέβη Άστον ε, σε απάντηση στην επιστολή της ε, πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο και λάβουμε υπόψη και το κόστος του να μην υπάρξει ένα επιχειρησιακό στρατηγείο. Υπάρχει επίσης το θέμα της ρήτρα της αμοιβαία συνδρομής που είναι και νομική υποχρέωση της συνθήκης και θα πρέπει να προχωρήσει και να την επεξεργαστούμε λίγο περαιτέρω. Υπάρχει και η συνθήκη της Γάνδης για τις στρατιωτικές δυνατότητες. Υπάρχει και η ομάδα για την πιθανή διαφοροποίηση ε, και να έχουμε αυτές τις battle groups οι οποίες θα είναι ένα μέσο που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετικές δομές ε, να χρησιμοποιούμε και τις ε, δυνατότητες ε, να έχουμε κάποιες μάχημες μονάδες που θα έχουν συμπληρωματικές ε, αρμοδιότητες και λίγο διαφορετικές από αυτές που είχαν καθοριστεί αρχικώς για τις μάθημες μονάδες. Υπάρχει το θέμα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Άμυνας και μέσω της αναγνώρισης των δύο βασικών οδηγιών που υπάρχουν για το θέμα αυτό. Κατόπιν, ίσως να μακρηγορώ βέβαια, eh, Υπάρχουν και κάποια επιπλέον κεφάλαια. Υπάρχει ένα κεφάλαιο εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια με κάποιες προτάσεις ε, πολύ συγκεκριμένες και να ενισχύσουμε τις συνέργειες μεταξύ των δύο πτυχών αυτών υπάρχει και μία, μία αναλυτική εξέταση των διαφόρων αποστολών και εξετάζουμε απλώς κάποια προβληματικά στοιχεία που προκύπτουν από τις αποστολές οι οποίες είναι εν με κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις ε, για κάποιες εξ αυτών ε, στη Βοσνία και σε κάποιες άλλες αλλά σας παραπέμπω στο γραπτό μου μνημείο και υπάρχει επίσης και μία μικρή ανάλυση για την ανάπτυξη των διαφόρων συμπράξεων, τους διαφόρους συνδηλαγόμενούς μας, το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση και τέλος τη συνεισφορά των τρίτων ε, χωρών στις διάφορες αποστολές. Αυτό είναι το περιεχόμενο σε γενικές γραμμές της έκθεσής μου. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψη των συναδέλφων και θα ήθελα να ακούσω και τις υποδείξεις τους και τις τροπολογίες τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ merci, monsieur. κύριε σα ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Τώρα θα κάνουμε μια κράψη ε, στις συνήθεις κανόνες λειτουργίας της ομάδας μας, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία συνάδελφό μας, η οποία θα πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ. Ε, θα σας ε, επενέσω και γενικά ήταν καλές οι διάφορες παράγραφοι. Παράγραφος 8 έως 39. Ε, Στην 45 ε, έως 453 ε, μιλάμε Η 47 είναι κάπως περίεργη, home και security. Για την αποστολή στο Κονγκό είστε λίγο επικριτική Τι εκεί ακριβώς είναι το θέμα. Στην 16 θα... έπρεπε να μιλάμε για το EUTM 60, 60. Η προηγούμενη ποια ήταν, 47. Και μετά 66. Ε, λίγο πιο ασθενή σε σχέση με το... την ασφάλεια. Και μετά δύο σημεία που νομίζω ότι λείπουν δεν έχουμε ανεξάρτητη ποιοτική αξιολόγηση των αποστολών. Και δεύτερον, μη εξάπλωση και αφοπλισμός. Ίσως και σε αυτό λίγο να συζητήσουμε. Αυτά, κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι εξαίρετη έκθεση. Έχετε πολλές παραγράφους για τις οποίες θα ήθελα να σας συγχαρώ. Merci, merci pour la brièveté de l'intervention. Είμαι πάρα πολύ για ήταν σύντομη. Ο αντιπρόεδρος του κ. Λίζικη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία στο Στασβούργο να συζητήσω με τον εισηγητή όσον αφορά το περιεχόμενο της εκθέσεως και είχαμε πρόβλημα με την κατανόηση ο ένας της γλώσσας του άλλου, είχαμε προβλήματα οργανωτικά. Πάντως, κατόπιν της αρχικής συζήτησης, διαπίστωσα την ουσία του κειμένου. Γενικά συμφωνώ. Πρόκειται για μια έκθεση αρκετά περίπλοκη. Ε, καταρχήν, με υπάρχουν βέβαια εδώ και εκεί κάποιες να μπορούμε να χτενίσουμε, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Ακριβώς να βρίσκουμε το πού επιδέχεται βελτίωση κάποιο κείμενο. Ο κ. επομένω επομένως, πάρα πολύ καλά δούλεψε Πρόκειται να υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες μέσα στην εβδομάδα. Γενικά το διεξιολογικό κείμενο. Θα συμπληρώσουμε κάποια σημεία, θα τα χτενίσουμε κάποια άλλα. Τα είπαμε την Κρυποπόψη όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών πληροφοριών και όσον αφορά την πρόσβαση ε, σε εμπιστευτικέ πληροφορίες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες ότι θα πρέπει να χρειάζεται όσον αφορά ε, τις υπηρεσίες μας που ασχολούνται με άμυνα και ασφάλεια. Επομένως, ε, ίσως θα πρέπει κάτι να προσθεθεί ε, ακριβώς όσον αφορά τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας. Επίση, όσον αφορά τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να έχουμε και σε αυτή τη διάταξη μια τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Κοπάκη το λόγο. Η έκθεση του συναδέλφου Γκουαλτιέρη παρουσιάζει με πλήρη και εξαντλητικό τρόπο τη συζήτηση η οποία πρέπει να διεξαχθεί σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας Τρία σημεία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά και αυτά θέλω να επισημάνω. Πρώτα απ' όλα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την παράγραφο 8 που τονίζει την ανάγκη για εσωτερική συνοχή και αλληλεγγύη παρόμοια με αυτή που επιτεύχθηκε μεταξύ των χωρών Σέγγεν. Θεωρώ ότι το παράδειγμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς η άμυνα σχετίζεται και με την έννοια των εξωτερικών συνόρων και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών Ωστόσο, ίσως θα έπρεπε να επισημανθεί πιο ξεκάθαρα η αντίφαση σε σχέση με την πραγματικότητα που παρά την ρήτρα αλληλεγγύη στη συνθήκη θέλει την κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας να περιορίζεται στις λεγόμενες αποστολές Πέτερσμπεργκ. Δεύτερο σημείο. Πολύ σωστά επισημαίνεται η ανάγκη δημοκρατικής νομιμοποίησης της πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας η οποία παραδοσιακά παραμένει στα ζητήματα που κυβερνήσεις προσπαθούν να κρατήσουν στη στενή σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους. Σε δύο σημεία στην έκθεση αναφέρεται ότι οι εκθέσεις και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ένα ακόμα σημείο όμως που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με την εξωτερική δράση αλλά και τους στόχους των ευρωπαϊκών αποστολών σε απόμακρα και επικίνδυνα μέρη του κόσμου. Τέλος, θέλω να συμφωνήσω σε σχέση με την κριτική που εκφράζει ο κύριος Γκουαλτιέρη στο σημείο 18 σύμφωνα με τα κενά που παρατηρήθηκαν στην προκαταρτική οργάνωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης σε σχέση με τη διαχείριση κρίσεων καθώς και την παράγραφο 21 σε σχέση με το Civilian Headline Goal, καθώς οι πολιτικές δυνατότητες δεν πρέπει να παραμελούνται και πρέπει να δούμε τη συνέχεια από εδώ και πέρα. Να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε δηλαδή κατά πόσο χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη, ίσως υπό τη μορφή ενός αναθεωρημένου Civilian Headline Goal που θα καλύψει τις ελλείψεις και θα εξασφαλίσει μια ισόρροπη ανάπτυξη πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων. Ε, θεωρώ επίσης για να κλείσω πολύ σημαντική την επισήμανση ότι χρειάζεται μία αναφορά στα μεγάλα γεγονότα της ε, Βόρειας Αφρικής. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν μια μεγάλη δοκιμασία στο επίπεδο της ασφάλειας, εσωτερικής και εξωτερικής, τόσο για τα κράτη του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνολικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια επισήμανση νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν όψη της παρένεσης σας στην αρχή σχεδόν ε, θέλησα να μην μιλήσω αλλά έχω κάποιες βασικές δυσκολίες με αυτήν την έκθεση, η οποία είναι πολύ όμορφα συνεταγμένη, όμως είναι μια άσκηση δημιουργίας ε, μύθων, ιδιαίτερα δαπανηρή. Και είναι και λίγο μεγάλη, πολλοί θα χαθούν εδώ μέσα νομίζω. Ίσως και αυτό να είναι κομμάτι του στόχου. Παράγραφος 3 μιλάει για τη στρατηγική αυτονομία στην ασφάλεια από ποιον θέλουμε αυτή την ε, στρατηγική αυτονομία. Αυτό φυσικά φαίνεται να υποστηρίζει όλο το επιχείρημα γιατί όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 3 ήδη γίνονται στο ΝΑΤΟ. Δεν κατάλαβα λοιπόν τη λογική. Να πάμε στην παράγραφο 74 Ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε για άλλη μια φορά τη λογική της παραγράφου, αν γνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτό. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιστροφή τη Γαλλία στην ολοκληρωμένη διοίκηση τη Ατλαντική Συμμαχία και θεωρεί ότι το γεγονό αυτό πρέπει να κάψει κάθε αντίσταση όσον αφορά στην ανάπτυξη μια κοινή αμυντική πολιτική. Δεν κατανοώ την λογική. Θεωρεί ότι πρέπει να ε, απαλλαγούμε οποιαδήποτε ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινή πολιτικής άμυνας. Επίσης, στο τέλος αναφέρεται και η ανάγκη να μιλήσουμε για τη Βόρεια Αφρική. Στην ουσία ε, προσυπογράφουμε την έκκληση της ε, δήλωσης ε, της Τρίπολης. Πολλά από αυτά που αναφέρονται εκεί στην παράγραφο 76 ίσως είναι πράγματα που τα έλεγε και ο κύριος Καντάφη. Ευχαριστώ, η κυρία Λουζίνγκ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ την ευχή του Προέδρου και να μην μπω σε αψημαχίες. Σε όλη την έκθεση Είχαμε ήδη συζητήσει κάποια πράγματα στην τελευταία συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η ομάδα μου δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως. Μόνο για την ε, γενική φιλοσοφία της ε, στρατιωτικής ε, πολιτικής άμυνας. Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία κριτικής στα οποία θα περιοριστώ. Στην παράγραφο 6 αναφέρεται ε, ότι υπάρχουν ε, αποστολές ε, στρατιωτικές και πολιτικές όχι μόνο στα πλαίσια της ΚΠΑ αλλά και για την προστασία από καταστροφές. Θεωρούμε ότι είναι λάθος η ΚΠΑ είναι ένα γενικό εργαλείο θα έλεγα. Θέλουμε ε, στρατηγικοποίηση της ε, αντιμετώπισης καταστροφών. Αυτό κάνουμε τουλάχιστον με το στρατιωτικό στοιχείο εδώ. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις που βλέπουμε από αυτόν τον περιορισμό. Στη παράγραφο 17 γράφεται από τη μία ότι υπάρχουν διαχωρισμούς μεταξύ της πολιτικής και στρατιωτικής ε, συνεργασίας. Όμως αυτό πρακτικά κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται. Το επόμενο θέμα είναι η παραγραφη 10, 11, 12 και κυρίως η 13 σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γράφεται πολύ συχνά για την έλλειψη του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά δεν βλέπω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η ομάδα μας ήδη έχει καταθέσει προτάσεις. Ε, Θα θέλαμε ο εθνικός έλεγχος στα κράτη-μέλη να ήταν καλύτερος και δεν θέλω να παρανοηθεί, όπως είπε και ο κύριος Μπροκ. Θέλουμε ένα, πλήρως, ένα πλήρες δικαίωμα πληροφόρησης, ακρόασης για τις αποστολές της ΚΠΑ, έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια, όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται, να μπορούν να ταξιδέψουν στους τόπους που υπάρχει στρατιωτική δράση. Επίσης για την διασφάλιση μιας κοινή δράσης ε, στην ε, συγχώνευση της ΚΕΠΑ και της ΚΠΑ με άλλες, ε, άλλους τομείς πολιτικής. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ποιες είναι οι προειδοποιήσεις των οργανισμών αναπτυξιακής βοήθειας προειδοποιούν για μια συνεργασία των στρατιωτικών και ανθρωπιστικών ε, αποστολών ε, θεωρούν ότι το να συγχωνεύσουμε στρατιωτικές και οικονομικές ε, αποστολές θα υπονόμευε ας πούμε τις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Τέλος, πολύ σοβαρή ε, κριτική θα ήθελα να ασκήσω στην ε, συνεχώς δομούμενη συνεργασία. Στην ε, παράγραφο 28 μιλάμε για μια υποχρέωση των κρατών μελών να ε, εξοπλιστούν και να δράσουν στρατιωτικά. Νομίζω ότι αυτό είναι κατά της δημοκρατίας. Αυτό δεν ε, υπονομεύει την, ε, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών σε επίπεδο στρατιωτικό και σε επίπεδο πολέμου. Και πώς τότε λέμε ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολιτικό χαρακτήρα. Για μένα η ειρήνη δεν ε, μπορεί να υπάρχει μέσα από στρατιωτικές προτεραιότητες. κοιτάξτε τι έγινε στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Σομαλία, στο Κονγκό. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν ε, τα επιχειρήματα αυτά ενισχύουν ακριβώς αυτό που θα θέλω να σας δείξω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήμουν από την αρχή. Νομίζω όταν ε, είναι κατά οι κομμουνιστές και ευρωσκεπτικιστές ε, αυτής της έκθεσης, τότε εγώ είμαι σε καλό δρόμο. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Η έκθεση είναι πολύ σημαντική γιατί η θέση του Κοινοβουλίου που εμείς εδώ στην Επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία έχουμε ε, βρει ε, είναι ότι θέλουμε να είναι αυτό ένα σημείο της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας. Είναι λοιπόν καλό το κείμενο με, με το κατάλληλο μήκο. Για την παράγραφο 34, για το κοινό στρατηγείο, επιχειρησιακό στρατηγείο, πρέπει λίγο να σκεφτούμε αν θέλουμε να ορίσουμε κάποιο χρονικό περιθώριο, να δώσουμε ένα, μια χρονική διάσταση. Ο συνάδελφος Φανόρντεν είπε και αυτός ότι είναι σημαντικό, όπως θεωρώ και εγώ, ότι ε, στην περίπτωση της Λιβύης οι Αμερικάνοι μας ρώτησαν ε, από ποιο αρχηγείο θα πρέπει να περιμένουν οι Αμερικάνοι ότι οι Ευρωπαίοι θα ε, αναλάβουν τις επιχειρησιακές και πολιτικές ευθύνες. Ζητούν να μάθουν λοιπόν από άποψη ΝΑΤΟ, από τους ε, Αμερικανούς τουλάχιστον συζητείται ξεκάθαρα αν μπορούμε να το κάνουμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ από την Τουρκία και να υπάρχει και μία έμεση αμερικανική συμμετοχή πολιτική ε, στη Βόρεια Αφρική, αν θα ήταν κάτι τέτοιο σόφρον. Αυτά σχετικά με το ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές ε, δομές. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε ε, μια χρονική διάσταση συγκεκριμένη σε αυτό το στοιχείο. Κάτι άλλο που πρέπει να δούμε αν θα συζητήσουμε είναι η σημασία της cyber security και του cyber war κυβέρνο χώρος, ε, πόλεμο στον κυβερνοχώρο και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η ε, Αμερικανική κυβέρνηση θέλει μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς στην Ευρώπη είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τις αντίστοιχες δομές και από την πλευρά της Αμερικής ξεκάθαρα αναφέρεται ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ της ασφάλειας στον στον κυβερνοχώρο σε πολιτικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Πρέπει εμείς να δούμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πώς θα ε, συνενώσουμε αυτά τα στοιχεία, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε για να είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν να προσθέσουμε μια παράγραφο για αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλή η έκθεση θεωρώ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ που ήσασταν πολύ συγκεκριμένος προς τα σημεία της έκθεσης που θέλατε να επικρίνετε. Κύριε Γκολτχέρη, μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτά, εάν θέλετε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα κάνω μια απόπειρα να απαντήσω επί της ουσίας, κυρίως για τα πιο συγκεκριμένα και πιο εύστοχα σχόλια και κατόπιν ε, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι για τα σχόλιά τους ε, ουσιαστικά μας ε, λένε ότι θα κάνουν και τροπολογίες, επομένως θα προσπαθήσω να σχολιάσω ως τροπολογίες. Για το σημείο 59 καταλαβαίνω τι ανησυχίε έχει ο κύριος Μπραντ, αλλά να σας επαναλάβω τι περιλαμβάνουν τα σημεία αυτά. Το θέμα της ε, διτής χρήσης και των δυνατοτήτων διτής χρήσης και το ρόλο στο πρόγραμμα πλαίσιο στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνα. Επομένως, ε, υπ' αυτήν την έννοια δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τώρα την ενίσχυση των παραγράφων 45 και 53 ε, που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θεωρούσα ως δεδομένο το γεγονός αυτό, διότι στην αρχή της ε, έκθεσης αναφέρω ότι επειδή ε, αλλάξαμε και δεν έχουμε πλέον δομή πυλώνων, όλες οι πολιτικές υποβάλλονται στις αρχές και τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλέον είναι δεσμευτικές. Η λογική λοιπόν της έκθεσης είναι να υποστηρίζουμε ότι ακόμα και από νομική ε, σκοπιά είναι πολύ πιο ισχυρός αυτός ο δεσμός από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την πτυχή αυτή στην ε, στις παραγράφους που αναφέρονται στη σχέση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, όπως έλεγε η κυρία Μπραντ. Τώρα, για την παράγραφο 47 και τον παραλληλισμό με την αμερικανική ε, εμπειρία μπορούμε με να τα διαγράψουμε αλλά δεν κάνω τον παραλληλισμό για να πω ότι θα πρέπει να μιμηθούμε αυτό το μοντέλο αλλά λέμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει κάνει κάποιες επιλογές οι οποίες ε, πλέον θεωρούν τη διάσταση της ασφάλειας μια, ασφάλ... Ε, μια διάσταση η οποία συνδέει πολύ στενά την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια και θεωρούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συντονιστεί με αυτή τη νέα διάρθρωση των πολιτικών. Η ασφάλεια στον κυρμένο χώρο, για παράδειγμα, η συζήτηση για τα SWIFT. Ε, είναι θέματα τα οποία κάπου στο δικό μας καταμερισμό εργασιών ε, φαίνονται ξεχωριστά στοιχεία της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, αλλά τελικώς είναι τμήμα μιας συλλογικής πολιτικής. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέλει να είναι πλήρως συνειδητοποιημένη ως προς αυτά που κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις για θέματα που αφορούν την ασφάλεια ξεχωριστά, χωρίς να συνδυάζονται οι συζητήσεις και να μην υπάρχει και πολιτική συζήτηση επί τα θέματος. Και επειδή το Κοινοβούλιο είναι ο χώρος διαλόγου μεταξύ της ε, πολιτικής ασφάλειας και ε, επίσης είναι και συνομοθέτης για την εσωτερική ασφάλεια, αλλά δεν είναι μόνο εσωτερική ασφάλεια, διότι το SWIFT δεν αποτελεί μόνο στοιχείο εσωτερικής ασφάλειας. Θεωρούμε ότι είναι το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αυτές τις διαστάσεις. Στόχο λοιπόν είχα να ενισχύσω το επιχείρημό μου με την παραπομπή στις ΗΠΑ, αλλά μπορώ και να το διαγράψω. Όσον αφορά τώρα την παράγραφο 60, Μισό λεπτό γιατί δεν θυμάμαι τι έλεγε. Υπήρχε το θέμα για τη Σομαλία. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια τροπολογία βελτίωσης. Στην παράγραφη 66 σαφώς μπορούμε να ενισχύσουμε λίγο τα στοιχεία αυτά. Θα δεχτώ τροπολογία που ενισχύει την διατύπωση της παραγράφου 66. Όσον αφορά τώρα την μη διάδοση όπλων και τον αφοπλισμό, αυτό το ανέφερα και στην αρχή πρόκειται για ένα τόσο περίπλοκο και τόσο ευρύ θέμα και προτίμησα να μην το αναφέρω και να μην έχω τη συνήθη παράγραφο που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, εάν οι συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να αναφέρονται, θα μπορούσα κάλλιστα να δεχτώ μια τροπολογία ή τροπολογίες για το θέμα αυτό. για τα σχόλια του κ. Λίζεκ, τον οποίο ευχαριστώ. Σίγουρα μπορούμε να ενισχύσουμε το θέμα της ε, υπηρεσίας πληροφοριών και της εργασίας του Situation Center και τις σχέσεις ε, με τις υπηρεσίες πληροφορίες. Άλλωστε σήμερα αναφερθήκαμε στο έλλειμμα πληροφοριών που έχουμε με τη Λιβύη Και στο θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ σίγουρα μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη διατύπωση. Ε, θα μπορούσαμε να δεχτούμε σχετική τροπολογία. Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε, όπως έλεγε η κυρία Κοπά, την ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης και προς τους πολίτες και τους εκπροσώπους των πολιτών, δηλαδή στα κοινοβούλια. Συμφωνώ επίσης και με τις άλλες προτάσεις της κυρίας Κοπά που αφορούν κάποιες άλλες παρατηρήσεις στις παραγράφους 18, 21 και στις, τα σχόλιά της για την Αφρική. Τα σχόλια του κυρίου Βανόρντεν συνάδουν ε, με αυτό το παγιωμένο όραμα που έχει για τον περιφερειακό ρόλο της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ο κύριος Βανόρντερ. Σεβαστά τα σχόλιά σας, δεν συμμερίζομαι τις απόψεις σας βέβαια. Και Είμαι υπέρ του, της πηγής έμπνευσης της έκθεσης που θεωρώ ότι είναι και η πηγή έμπνευσης ε, της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου αλλά και της συνθήκης της ΟΒΑΝΑς ε, την οποία υπέγραψαν και κύρωσαν και οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις σας ε, για την παράγραφο 74, αν δεν κάνω λάθος, εγώ θεωρώ ότι η επιστροφή της Γαλλίας ε, στην ολοκληρωμένη διοίκηση του ΝΑΤΟ μπορεί να διασκεδάσει και τις υποψίες μια αντίφασης μεταξύ μιας ευρωπαϊκής ανάπτυξης άμυνας και του ΝΑΤΟ θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να είναι ευνοϊκό και να ευνοήσει και τη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Η διακήρυξη της Τρίπολης καταλαβαίνω ότι στις μέρες που βιώνουμε το να αναφέρεται κάποιο στη διακήρυξη της Τρίπολης μόνο υποψίε μπορεί να δημιουργήσει, αλλά είναι το σημείο στο οποίο έγινε η Σύνοδος Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και την υπέγραψε η ε, προεδρεύουσα νομίζω το Μαλάου είχε την προεδρία τότε της Αφρικανικής Ένωσης και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος Φαν Ρόμπαϊ και αναφέρεται και λέει πράγματα και τα οποία δυστυχώς παρά το γεγονός ότι υπεγράφησαν στην Τρίπολη είναι πράγματα τα οποία συμμεριζόμαστε όλοι. Δεν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μην αναγνωρίζουμε ότι επί της ουσίας τα σημεία στα οποία η Αφρικανική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λιβύη συμφώνησαν είναι σημεία τα οποία αφορούν τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής για την ασφάλεια και είναι πράγματα τα οποία μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Είναι στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν με θετικό τρόπο και στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε νομίζω το Δεκέμβριο για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις της συναδέλφου Λούζινγκ και αυτές ε, συνάδουν με τις απόψεις της και πάλι διαφωνώ μαζί της. Οι πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις σας ε, γεννούνται από αυτή τη διαφορετική τοποθέτηση που έχετε. Δεν θεωρώ ότι με σοκάρει μία παράγραφος ε, η οποία αναφέρεται σε ένα άρθρο της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ε, μόνιμη διαρθρωμένη δομή. Σε καμία περίπτωση αυτό το άρθρο δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη να κάνουν τη δική τους πολιτική, αλλά είναι μία διάταξη η οποία ίσως προβλέπει ένα πιθανό μέσο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να καθησυχάσω λοιπόν την κυρία Λούζινγκ. Δεν υπάρχουν ε, υφέρπουσες ε, επιπλοκές ε, με τη δημιουργία μιας μόνιμης δομής. Σε πιο γενικές γραμμές τώρα να πω ότι θεωρώ ότι ε, ο προεξάρχον ρόλος της ευρωπαϊκής μεθόδου, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ε, πολιτικές ε, που έχουμε για τα θέματα αυτά και μας κάνουν περήφανος που είμαστε Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι, δεν αντιφάσκουμε το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες στρατιωτικές δυνατότητες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για το σεβαστό του διεθνούς δικαίου και των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο και πιο συνολικό τρόπο την πρόκληση ε, του να είμαστε αξιόπιστοι παράγοντες στον ε, σημερινό κόσμο. Τέλος, τα σχόλια του κυρίου Έλερ. Με βρίσκουν σύμφωνο. Τον ευχαριστώ και για τα θετικά σχόλια που έκανα για την έκθεση. Άλλωστε η έκθεσή μου ε, αναζωογονήθηκε πολύ και από τα επικοδομητικά του σχόλια και επομένως μπορεί να χαίρεται που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της ε, έκθεσής του για το συγκεκριμένο θέμα σχέσης πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους. Συμφωνώ για την ε, προθεσμία για το επιχειρησιακό στρατηγείο και νομίζω ότι το παράδειγμα το οποίο έκανε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καταδεικνύει ακριβώς ποια είναι η γενική φιλοσοφία της έκθεσής μου και ποια είναι αυτή η ανάγκη να συνδυάσουμε διαφορετικές διαστάσεις προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική πολιτική συνοχή. Το παράδειγμα που μας έκανε είναι χρήσιμο και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Bien, merci beaucoup. Μάλιστα, λέω πρώτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας υπενθυμίζω. Τροπολογίες καλή την ημερομηνία 8η Τρίτου και επόμενη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις 15 Μαρτίου κατόπιν της ακροάσεως για την ε, αποστολή στην Βοσνία. Και τώρα προχωρούμε ή στην έκθεση. όσον αφορά μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία οποία προσφέρεται από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγης προέκυψε από το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Τον Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε τις προτάσεις της στην Επιτροπή μας. Και έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον προηγούμενο μήνα, όχι συγγνώμη, συγγνώμη, ο πρόεδρος, αρχάς Φεβρουαρίου όσον αφορά τις προτάσεις. Η κυρία Κοπά μας ε, ανέφερε τα βασικά σημεία της ε, εκθεσής της, ε, πολιτικές ομάδες τοποθετήθηκαν και έχουμε 29 τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Και έχουμε τις ήδη 15 τροπολογίες οι οποίες προτίθενται εκεί από την, την συγκίτρια που θα δώσω τώρα Τράτη κοιτάζει την κυρία Κοπά για να μας παρουσιάσει τις αλλαγές και κατόπιν θα συζητήσουμε για τους κύριους uh, first... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που θεωρώ πάρα πολύ σημαντική βοήθεια και συμβολή διότι πρόκειται για κάποια έκθεση ε, τεχνοκρατική, τεχνική και όχι ιδιαίτερως εύκολη. Οπότε ευχαριστώ και την κυρία Ροντόβα για τη συνεργασία της και γιατί απεδεχθεί το να έχουμε έναν κέντρο κατευθυνόμενο έλεγχο για την υλοποίηση και εφαρμογή των βασικών προτύπων όσον αφορά για αυτές τις ε, κυβερνητικέ υπηρεσίε. Όπω είδατε, έχουμε εδώ πέρα κάποιε κοινέ τροπολογίε και έτσι θα δούμε ε, το, το, πώ θα έχουμε στο κέντρο του συστήματο την Κομισιόν και θα υποπτεύει και θα λαμβάνει κάποια θετικά μέτρα ε, σε περίπτωση κάποιου είδου παραβίαση των όσων προβλέπει ο οργανισμό τα κρατημέλη πλευρά του πρόκειται να έχουν την αρμοδιότητα τη εφαρμογή και τη στηρίσεω των εθνικών διατάξεων, ε, που σύμφωνα με τον κανονισμό. Πέραν αυτών ε, θα πρέπει να δούμε το κατά πόσο δεν θα υπάρχει κάποιο είδους ε, ρίσκο και πώς δεν θα έχουμε κάποιο είδους παραδείσων διατάξεων για την διοδότηση και επίσης θα μπορεί κανείς να προσφύγει για οποιαδήποτε απόφαση που θεωρεί ότι είναι αβάσιμη. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους εποπτεία, κάποιο είδους σύστημα κυρώσεων σε δύο βαθμούς ή σε δύο επίπεδα, ε, κρατικό και ενωσιακό. Και θα προσπαθήσουμε επομένω να καλύψουμε οποιοδήποτε θεμητό αίτημα των εμπλεκομένων. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι έτσι θα είναι η εφαρμογή πιο ε, ισορροπημένη όσον αφορά την επικουρικότητα. Και άλλωστε η αρχική μου πρόθεση αυτή ήταν. Τώρα, σύμφωνα τι άλλε ε, τροπολογίε, όπω σα είπα, οι περισσότερε ε, βοηθούν ώστε να καταλήξουν σε μια <clears throat> θετική ε, έκθεση της Επιτροπής μας. Τώρα θα σας πω για ποιε δεν συμφωνώ, για ποιε έχω κάποιες επιφυλάξεις και θέλω να τις συζητήσουμε. Ξεκινώ με της κυρίας Ρέτοβε, την υπεροπολογή 14 ή 40, 40, 40 διευθυντής που αφορά την χρηματοδότηση του συστήματος και επίσης προτείνει το, το πώς θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το PRS, να, τι, τι, τι PRS να την ε, τρέξει. Ε, δεν έχω τίποτα να προτείνω, δεν, θέλω να πω τίποτα ε, του κατά πόσο χρειάζεται ε, κάποιο είδου χωριστή δομή, χωριστή χρηματοδότηση για την PRS. Νομίζω όμως ότι κατά τη γνώμη μου αυτή η τροπολογία υπερβαίνει τις αρμοδιότητές μας και επομένω προτείνω να μην την εγκρίνουμε. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Λούζιν και τι δικέ τροπολογίε, δυστυχώ δεν μπορώ να δεχθώ την υπαρτιμόνα 17, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένω έχει ισχυριστεί ότι το Γαλιλαίο είναι αξιόλογο σύστημα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των αποστολών της και Όμως συμφωνώ με την υπαριθμόν 42 τροπολογία της συναδέλφου γιατί ε, συνάδει προς τα όσα προσβεί το Κοινοβούλιο και οι συνδίκτες Λισαβόνας προβλέπουν υπάρχει κάποιο είδου στάνταρ παράταση, ε, επιμήκυνση των σχετικών χρονικών διαστημάτων. Τώρα, κύριε Γιατιμάκη, ε, έχουμε πρόβλημα μόνο με την υπαρχμόνη 26. Δεν ενδέχομαι, διότι σημαίνει ότι θα πρέπει να απαλληφθεί η διάταξη που λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο όποτε υπάρχει κάποιο θέμα. Τώρα, κατόπιν ε, των τροπολογιών Μπουτικόφερ, οφείλω να σας πω ότι η τροπολογία του 16, 18, 19 και 22 επισημάνουν κάποια σημαντικά ζητήματα, δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Όμως διατηρώ κάποιες ε, επιφυλάξεις για το κατά πόσον αυτός ο κανονισμός είναι το, το, πιο κατάλληλο μέσο. Η 18 επίσης νομίζω ότι συνάδει προς τον υπόλοιπο κανονισμό. Σύμφωνο με την τροπολογία. Πρόκειται άλλωστε για κάτι το οποίο και εγώ το είχα πει ως αυτή τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των προγραμμάτων ε, ε, δορυφικής ραδιοπλοήγησης με το 19 όμω δεν συμφωνώ. Δεν είναι σωστό να αναφέρουμε συγκεκριμένε χώρε. Όσον αφορά τι άλλε τροπολογίε, ε, είναι κάτι σαν ε, πολιτικέ δηλώσει, Δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να καλυφθούν με ένα νομικό κείμενο όπω αυτό ο κανονισμό. Πάντως είδα ότι ο κύριος ε, Λαμπέρτ επίση έχει ε, κάποιες σαν κάτι που θα μπορούσε να επισυναυθεί ως παράρτημα. Ίσως αυτή είναι μια δόκιμη λύση. Τη θεωρώ λογική. Και επίση θέλω να ρωτήσω τους αδέλφου ε, κατά πόσο μπορούν να συμφωνήσουν για μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Ρόιτοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα εγώ θα ήθελα να συμφωνήσουμε την έκθεση. Συμφωνώ με όσα είπε η κυρία Κόπα. Επίσης ε, σας ευχαριστώ ε, και χαίρομαι για το ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάτι όσον αφορά τις υποχρεωτικές κυρώσεις. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιες κυρώσεις που είναι μεν αγώγιμες κατά κάποιο τρόπο, επιβάλλονται από κάποιο δικαστικό όργανο, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι εφικτό νομικά να επιβάλλουμε το πρόστιμα και επίσης ιδίως όσον αφορά την ε, άρση της ε, άδεια λειτουργίας. Επίσης ε, συμφωνώ σε όσα το Κοινοβούλιο έχει πάντοτε προωθήσει σαν λύσεις κυρίως για τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας ή όσον αφορά το άρθρο 4, όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Επίση, θα πρέπει να γίνονται κάποιοι περιοδικοί έλεγχοι και θα πρέπει αυτό να προβλέπεται από το σώμα του κανονισμού. Αυτά είναι σημαντικά σημεία και εγώ διατηρώ κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά τι τροπολογίε 6 και 8. Εγώ θα ήθελα να τα συζητήσουμε αυτά τα δύο σημεία. Το άρθρο 2 λέει για τα κράτη-μέλη που έχουν την PRS και ότι δεν υπάρχει περιορισμός σε συγκεκριμένες χώρες νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε όψη ποιες χώρες έχουν προβλέψει έχουν ζητήσει την πρόσβαση να γίνει ρύθμιση με χωριστή παράγραφο. Τώρα, το, το θέμα της χρηματοδότησης δεν έχει ξεκαθαριστεί Νομίζω ότι για όλες τις χώρες θα πρέπει ό,τι θεσπιστεί να είναι δεσμευτικό. Και δεν ξέρω η συγγήτρια τι λέει όσον αφορά τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στο άρθρο 2. Θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές ή όχι. Τι γίνεται και με το άρθρο 8, την τροπολογία δηλαδή του άρθρου 8, γιατί εκεί λέει ότι οι χρήστες μπορεί να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Και όσον αφορά τους χρήστες του, της PRS ή μιλά για χρήστες δεκτών του PRS. Λέμε εδώ πέρα για νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, όμως τι γίνεται με κυβερνητικά οργάνα και αυτά δεν είναι ε, νομικά πρόσωπα. Εγώ σας τονίζω ότι θα πρέπει και τα κυβερνητικά όργανα, κυβερνητικές υπηρεσίες να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να καταστούν χρήστες του συστήματος. Φυσικά και νομικά εδώ υπάρχει πιο πρόβλημα να βρούμε κάποια λύση. Και να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση σύντονη με τα όσα ήδη προβλέπονται. Κάπως να δούμε τι θα κάνουμε για να καλύψουμε και τις κυβερνητικές υπηρεσίε. Να, μια λύση που θα μπορούσε να δοθεί στο πρόβλημα. Επίσης, έχω ένα άλλο πρόβλημα και έχω να σας προτείνω κάτι. Για το άρθρο 10. Λέμε για τις τρίτες χώρες που και αυτές θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, σε αυτό το, το, το, τον έλεγχο να, να πρέπει να υπαχθούν. Όμως εγώ να σας πω ότι στην τροπολογία 40 μνημονεύεται υπόθεση χρηματοδότηση για τις υπηρεσίε PRS. Εδώ έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις και δεν ξέρω μέχρι ποιου σημείου η εισηγήτρια εδώ ε, είναι 100% εύστοχη. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα στην Επιτροπή μας. Να μην αποτελέσει πρόβλημα. Να, να βρούμε κάποια συνεπική λύση. Και η τροπολογία αυτή να προωθηθεί και η Επιτροπή να βρει κάποια λύση. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στην αρχή της διαδρομής όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό. Πάντως έχουμε και κάποιες άλλες τροπολογίες που αφορούν κυρίως τη γλωσσική διατύπωση, κυρίως όσον αφορά την τσεχική εκδοχή του κειμένου, που υπάρχουν και καλύτερες διατυπώσεις, επίσης συμφωνώ με τις τροπολογίες των φιλελευθέρων. Εκεί που ζητείτε να ρυθμιστεί περισσότερο λεπτομερώς η πρόσβαση. Να σας πω τις προτάσεις μου και γράφος γιατί νομίζω ότι η υποχρέωση πληροφόρησης και ενημέρωση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να κατοχυρωθεί και να βελτιωθεί με αυτόν τον τρόπο το υπαρχόν σύστημα και η δυνατότητα πρόσβασης. Λείπει μία τέτοια ρύθμιση. Το να μπορεί το Κοινοβούλιο έτσι να έχει τον εκτενέστο δυνατό έλεγχο. Επίσης δεν συμφωνώ Η την τροπολογία που λέει ότι το σύστημα δεν θα χρησιμοποιείται για τα όπλα. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Βουτικόφερ. Εκεί που είπαμε για την τροπολογία 16 εκεί που είπαμε ότι δεν είναι πάρα πολύ εντελική η ρύθμιση όσον αφορά την χρήση για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρα λέμε ότι για οπλικά συστήματα θα ισχύει η ρύθμιση. Οπότε και συμπληρωτώ το κείμενο. Και συμφωνώ επομένω με την ε, εισηγήτρια. Καλά, περισσότερο ιδεολογικό είναι το θέμα και κάποιες χώρες θεωρούν ότι πάνω σημείο και μετά οι ρυθμίσεις αυτές ξεπερνάνε τον σκοπό της σύνταξης του κανονισμού. Θα βάλω εδώ τελεία, αλλά πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν συμφωνώ να πούμε για στρατό να πούμε ότι δεν θέλουμε σε στρατιωτική χρήση. Αυτό ναι, είναι σωστό. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή, κύριο Κίλμαν. Ευχαριστώ. Να πω ότι διάβασα τις τροπολογίες με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ε, και τα σχόλια που έγιναν για αυτό το θέμα στην εισηγήτρια. Νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που έχουν πιο πολύ δηλωτική φύση. Αναρωτιέμαι αν κάποιες θα μπορούν να αναφερθούν στα εκτιμώντας ε, και στις αιτιολογικές θέσεις ειδικότερα για τα στρατιωτικά, να αναφερθώ στο ψήφισμα που έχει ήδη εγκρίνει η Επιτροπή αυτή. Δεν είναι κάτι καινούριο λοιπόν. Απλώς να πω ότι το PRS είναι ένα από τα μία από τις πέντε υπηρεσίες του συστήματος Γαλιλαίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και νομίζω ότι έχουμε βρει ε, το διαχωρισμό μεταξύ των κοινών ελάχιστων στάνταρ που πρέπει να γίνουν σεβαστά από τα κράτη-μέλη και μετά ε, στην κυριαρχία των κρατών μελών το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση τις αρμοδιότητές τους, τις δυνατότητές τους υπό τον έλεγχο της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τέλος, ε, νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λιγάκι κατά κάποιο τρόπο όταν μιλάμε για τον κανονισμό 683 ε, που θεσπίζει το σύστημα του 2008 και δίνει ξεκάθαρο ρόλο στην Επιτροπή και στο GSA. Άκουσα από πολλούς να λένε ότι θέλουν περισσότερες αρμοδιότητες στο GSA. Νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο αυτά που αποφασίσαμε το 2008. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτε θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα πω ότι δεν συμφωνώ, το ΕΛΚ δηλαδή, δεν συμφωνεί με την πρόταση της κυρίας Λέσινγκ που λέει ότι ο Γαλιλαίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ε, δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση που έγινε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, κάποια απορία σχετικά με το ότι θεωρείτε εσείς και την κυρία Λουζίνκ. Δεν είναι καινούργια συζήτηση, κυρία Κοπά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν σχεδόν ε, το πιο σημαντικό πράγμα που είπατε, γιατί ε, κατά κάποιο τρόπο είχα αρχίσει να μπερδεύομαι. Σας ευχαριστώ πολύ να δώσω μία-δύο σύντομες απαντήσεις σε κάποια από τα σημεία της κυρίας Ρόιτμπερτ για την τροπολογία 6 καταρχάς. Νομίζω ότι η τροπολογία αυτή δεν θέλει να αλλάξει την αρχή ότι μόνο τα κράτη-μέλη που θέλουν να επωφεληθούν και θα παρέχουν στο σύστημα θα έχουν απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση. Όσοι θέλουν λοιπόν να συμμετάσχουν μπορούν να έχουν αυτή την πρόσβαση. Αν θεωρείτε όμως ότι δεν είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα επαναδιατύπωσης. Αυτό ήταν απλά ένας τρόπος για να δώσω τη βασική αρχή. Τώρα για την τροπολογία 8. Η δική μου τροπολογία ήθελα να τονίσω ότι τους κυβερνητικούς φορείς γιατί νομίζω ότι Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι διάφοροι τομεί ε, της κυβέρνησης, της διοίκησης των κρατών μελών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως το σύστημα. Τίποτα παραπάνω λοιπόν, δεν προσθέτω κάτι, απλά δίνω έμφαση στο θέμα αυτό. Σχετικά με τη χρηματοδότηση, φυσικά είναι σημαντική, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή είναι η σωστή γνωμοδότηση για να μπορέσει αυτό να αναλυθεί. Δεν θα μ' άρεσε πολύ να το έχω στο κείμενο. Ε, αποδέχομαι την προφορική σας ε, τροπολογία σχετικά με τις πληροφορίες όταν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, όταν καταστραφεί το σύστημα. Ε, σκέφτομαι επίσης να καταθέσω τρεις προφορικές τροπολογίες προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να βρω ένα συμβιβασμό για το κείμενο. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα σας στείλω τις επόμενες ημέρες λοιπόν τις προτάσεις μου για τις προφορικές τροπολογίες όπου θα τονίζω ότι είναι μια τεχνολογία διτής χρήσης. Εργαζόμαστε επί αυτής της βάσεως, αυτό είναι το σημαντικό. Και φυσικά εδώ σε αυτή την αίθουσα ακούγονται οι διάφορες απόψεις, όμως για την ομάδα μου και για το ΕΛΚΑ είναι πολύ ξεκάθαρο και έτσι δουλεύουμε. Αυτά νομίζω ότι ήθελα να τονίσω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σέλλερ. Μια ε, παρατήρηση για το στοιχημείο 7 της της διάταξης. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο υπάρχει άλλη παρέμβαση. Όχι, το επόμενο βήμα λοιπόν θα είναι στην αφέτη ψηφοφορία στις 10 Μαρτίου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα μας μένουν τα διάφορα που θέλετε να θίξετε πριν λήξουμε τη συνεδρίαση, κύριε Έλλερ. Δύο σημεία Ξέρουμε ότι η υπηρεσία έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να μεταφράζει σε διάφορες ε, γλώσσες. Ε, να πω απλώς ότι στην έκθεση του κυρίου Γκολτιέρη στα γερμανικά υπάρχουν γραμματικά και άλλα τέτοια λάθη. Ξέρω ότι είναι τα γερμανικά δύσκολη ε, πρόταση, ε, γλώσσα, αλλά ας βάζουμε ένα ρήμα στην πρόταση για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Επίσης ήθελα να δω αν θα μπει στην ημερήσια διάταξη, αν το σκεφτόμαστε, να υπάρξει μια γνωμοδότηση, μια θέση σχετικά με την ε, έκθεση για την ασφάλεια στην Επιτροπή Ήτρε. Μιλάμε για τις ε, στρατιωτικές ε, και ε, διαστάσεις και τις διαστάσεις ασφαλείας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά να λάβουμε θέση και για αυτό το θέμα. Les deux points sont, sont justes et, bien notés pour... Euh, και τα αιτήματα και τα σημειώνουμε. Για το δεύτερο θέμα σας, για την γνωμοδότηση η απόφαση λαμβάνεται σε επίπεδο ΑΦΕΤ. Έχουμε υποβάλει την πρόταση στο Προεδρείο της ΑΦΕΤ, λοιπόν, στους συντονιστές. Περιμένουμε την απάντησή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Στις 15 Μαρτίου το επόμενο ραντεβού μας ε, για λέξικο ψηφοπαίδιο. έχω ε, Χωσιφοπέδιο για Βοσνία και νέα έκθεση Γκολτιέρη. Ευχαριστώ.